Uh, uh, λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο πάνελ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ξεκινάει τώρα η μετάδοση μέσω διαδικτύου της εκδήλωσης. Από εδώ και πέρα λοιπόν μεταδίδεται ζωντανά παγκοσμίως. Καλωσορίζουμε λοιπόν και το διαδικτυακό κοινό μας πλέον ε, στο σεμινάριο αυτό για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ασύλου και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι από τούτο και στο εξή οι συζητήσεις ε, πλέον καταγράφονται ε, σε αντίθεση με το προηγούμενο πάνελ που ήταν άτυπη συζήτηση. Έχουμε δύο προσκεκλημένους λοιπόν εδώ οι οποίε θα μας δώσουν την άποψη πλέον της πρώτης γραμμής. Εκ δεξιών έχουμε τη Μελίτα Σούνιτς, η οποία είναι εκπρόσωπος και ε, υπάλληλο ε, των Περιφερειακών Εξωτερικών Σχέσεων του ε, UNHCR, της ε, Υπηρεσίας Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών και εξ αριστερών η Άννα Λόπεθ Φοντάλ, η οποία είναι υπεύθυνη τύπου και ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θέματα προσφύγων και και Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στις ομιλήτριες ε, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας γύρος ερωταποκρίσεων. Θα ήθελα να ζητήσω να <laughs> σεβαστείτε τους κανόνες λοιπόν και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ο λόγος στη Μελίτα Σούνιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μαζί σα. Συνήθω αυτό λένε συνήθω οι ομιλητέ στην πρώτη πρόταση και στη συνέχεια αρχίζουν να μιλούν ε, ε να σταματούν. Δύο λόγια λοιπόν θα πω. Ο Ιταλός συνάδελφος που δυστυχώ που διαφεύγει το όνομά του έθεσε μια τελευταία ερώτηση για τι ε, δυσκολίε κατανόηση τη ε, νομοθεσία για το άσυλο και αυτό με οδηγήσει σε αυτό που θέλω να σα πω. Η νομοθεσία για το άσυλο σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα προηγμένη, πολύ εξελιγμένη. Ε, είναι ένα σύνολο κανόνων ε, που εξελίσσονται συνεχών και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς ε, έχουμε σκοπό από πλευράς UNHCR να ετοιμάσουμε ένα φυλάδιο που θα εξηγήσει σε εσά σε τι αναφέρονται οι νομικοί και όλοι όσοι ασχολούνται με το άσυλο και από εκεί και πέρα θα επαφίεται στις διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με το άσυλο και ε, στη UNHCR και στις εθνικές κυβερνήσεις να τα μεταφράσουν σε πιο απλή γλώσσα ώστε να είναι κατανοητά ε, και να μπορούν να τα κατανοήσουν και ετούντες άσυλο, επομένως να βρίσκονται και στη γλώσσα τους. Ε, θα ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για την γενικότερη εικόνα. Να ξεκινήσω από τα θετικά στοιχεία. Η Ευρώπη, η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο μεγαλύτερος χώρος που διαθέτει τόσο εξελιγμένο και ε, ανεπτυγμένο σύστημα ασύλου παγκοσμίω. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή στον κόσμο ώστε να υπάρχουν τόσο πολλοί κυβερνητικοί φορεί, δικηγόροι, μη κυβερνητικέ οργανώσει και δημοσιογράφοι που να ασχολούνται με το ζήτημα, να το κατανοούν και να στηρίζουν την έννοια του ασύλου και την έννοια τη προστασία σε ανθρώπου που χρειάζονται προστασία. Αυτά είναι τα θετικά. Και πάλι θετικό είναι το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί ιδιαίτερη πρόοδος ε, για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με εναρμονισμένη προσέγγιση, το οποίο υποστηρίζουμε και εμείς ως Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών εδώ και καιρό και δίνουμε και πολλές ε, συνεισφορές για την εκπόνηση της νομοθεσίας όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Και να αναφέρω ότι η Ευρώπη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως κάθε κράτος μέλος είναι από τους μεγαλύτερους εισφορείς ε, για την στήριξη διεθνών ανθρωπιστικών κρίσεων και για τις εσωτερικές κρίσεων, ε, κρίσεις προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός, αλλά αν προσθέσουμε και τη συνεισφορά των κρατών μελών, θα δείτε ότι οι Ευρωπαίοι πραγματικά υποστηρίζουν το άσυλο. Αυτό ήταν το θετικό, δυστυχώ πρέπει να σας πω και τα αρνητικά. Ε, σύντομα θα έχουμε και επί χάρτου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σύλλου. Ε, προσπαθούμε να επηρεάσουμε όσο το περισσότερο μπορούμε, επειδή είμαστε και αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ε, Σύμβασης Προσφύγων της Γενέβης του 1951 και ε, προσπαθούμε ακόμα να επηρεάσουμε και κάποια από τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί ακόμα, όπως για παράδειγμα το Eurodac, με ποιο τρόπο θα ε, δίνονται αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα στην αστυνομία, τι γίνεται όταν έχουμε να κάνουμε με βάλωτα άτομα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και συνόδευτων ανηλίκων. Προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή να βοηθήσουμε να τελειοποιηθεί αυτό το πολύ μεγάλο πακέτο νόμων για το άσυλο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για να προστατεύει τους πρόσφυγες. Όμως, στο τέλος θα έχουμε πάρα πολλά χαρτιά, χαρτούρα. Από τη χαρτούρα βέβαια στη ζωή καταλαβαίνουμε ότι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και επειδή είχαμε ανέκαθεν οδηγίες για το άσυλο, δεν είναι κάτι καινοφανές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε όμως τι γίνεται με την εφαρμογή, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές. Αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών που έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης. Η Σλοβενία, νομίζω, και η Ιρλανδία, κάποιες χώρες της Βαλτικής. Ε, και έχουμε και χώρες στις οποίες ε, υπάρχει πραγματικά σοβαρή πιθανότητα να σας ε, αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα και να υπάρχει προστασία. Και ακόμα και αν δείτε και τις ίδιες ομάδες ανθρώπων, Αφγανοί ή Σύροι. σε κάποιες χώρες θα τύχουν προστασία, σε κάποιες άλλες όχι. Επομένως, ε, ε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ε, τα εφαρμόσουμε αυτά στην πράξη και δυστυχώς από το χαρτί στην πράξη υπάρχει ένα χάσμα. Και εμείς ως ενδιαφορεωμένοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε, αλλά και εσείς ως δημοσιογράφοι πρέπει αυτό το τεράστιο νομικό επίτευγμα να προσπαθήσουμε να του προσδώσουμε ζωή και να βοηθήσει πραγματικά τους πρόσφυγες. Ε, τι είναι αυτό το οποίο όμως υποκινεί την νομοθεσία ασύλου. Ε, καταρχάς ε, έχουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφενός που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και τις χώρες οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική τους νομοθεσία. Από εκεί και πέρα έχουμε τις εθνικές κυβερνήσεις, από εκεί και πέρα τα ανώτατα δικαστήρια και τα εθνικά ανώτατα δικαστήρια, αλλά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν λάβει αποφάσεις οι οποίες αποτέλεσαν ορόσημο στο παρελθόν και μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και από εκεί και πέρα υπάρχει κοινή γνώμη και οι εθνικέ κυβερνήσει, οι οποίε εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ε, την, το τι γίνεται και ξέρετε ότι η κοινή γνώμη ορισμένε φορές μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις πάρα πολύ. Κάποιοι λένε ότι αυξάνεται η ξενοφοβία και τα πράγματα χειροτερεύουν συνεχώς. Εγώ δεν θα ήθελα να τα βλέπω όλα υπό αυτό το πρίσμα. Αν ε, ανατρέξουμε στο τι συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια, το πώς αντιλαμβανόμασταν το άσυλο τότε και πώς το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, έχουν ε, σίγουρα επιδεινωθεί τα πράγματα. Από την άλλη όμως πολύ συχνά διαπιστώνω και είμαι βέβαιη ότι και εσείς μπορεί να έχετε αντίστοιχα παραδείγματα στις χώρες σας ότι ξαφνικά υπάρχουν κάποιες ασυνήθιστες συμμαχίες, διότι ε, θα απελαθεί ο τάδε και ένα ολόκληρο χωριό ή μια ολόκληρη πόλη, ένα ολόκληρο σχολείο του στηρίζει. Οι εφημερίδες ε, συνεχίζουν να γράφουν για αυτούς τους αλλοδαπούς και το πώς ε, δυνατούν να ενσωματωθούν και ξαφνικά στηρίζουν τον συγκεκριμένο. Δεν είναι λοιπόν φθήνουσα η πορεία στην πραγματικότητα, είναι ένα σκαμπανέβασμα και το βλέπουμε αυτό και στις εφημερίδες και στη δημόσια συζήτηση που γίνεται σε διάφορες χώρες, ακόμα και στη δημόσια συζήτηση των ε, ανθρώπων που συνήθως είναι ύποπτοι, ακροδεξιά κόμματα που χρησιμοποιούν το αίσθημα ξενοφοβίας και το φόβο για τους αλλοδαπούς ε, στην ε, δημόσια συζήτηση. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχουν διακυμάνσεις, δεν είναι παντού σε αύξηση, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το ομολογώ, αλλά ε, σε κάποιες χώρες έχει μειωθεί η τάση ε, και έχω ε, ακούσει και τις καλύτερες και τις χειρότερες συζητήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας και εδώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και μία συζήτηση. Πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση όπου υπάρχουν τα μέσα, έχουν αναπτυχθεί, υπάρχουν, πρέπει να εφαρμοστούν και οι χώρες πλέον έχουν χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να τα εντάξουν στην εθνική τους νομοθεσία και να τα εφαρμόσουν. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς από κοινού να ε, υποστηρίξουμε όλη αυτή την πορεία και η συζήτηση ή μάλλον να σας το θέσω αλλιώς η συζήτηση είναι αρνητική όταν συζητάμε μόνο για κανόνες, κανονισμούς και στατιστικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή αρχίσουμε να αναφερόμαστε στους ανθρώπους, στη μοίρα τους. Αλλάζουν τα πράγματα και ακόμα και στο, στα ίδια μέσα ενημέρωση, στην ίδια τηλεόραση, στην ίδια εφημερίδα θα δείτε μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Και εδώ νομίζω ε, ότι είναι ο δικός μας ο ρόλος, πρέπει να ξαναλήξει η συζήτηση, να πούμε ότι ναι, έχουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την προστασία τους. Δεν υπάρχει μία και μόνο ομάδα και με αυτό ολοκληρώνω η τελευταία μου φράση που να μην έχει βιώσει τόσο πολύ δραματική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν ε, τόσο δύσκολες συνθήκες ως πρόσφυγες ανά τον κόσμο και αν θέλουμε να τους στηρίξουμε, αν θέλει η Ευρώπη να ε, ε, φανεί αντάξια των ιδανικών της, τα οποία ξεκινούν και από τη Γαλλική Επανάσταση και ακόμα πιο πριν, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, το αγάπα των πλησίων σου, ανάλογα με το πώς το αποκαλείτε με βάση τις ιδεολογικές σας πεπιθήσεις, θα πρέπει να ε, προσδώσουμε ζωή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Σύλλου και αυτό θέλω να συζητήσω μαζί σας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ, πολύ Μελίτα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην δεύτερη συγγετριά μας, την Άννα Λόπες. Κράτησε την υπόσχεσή σου, Μελίτα. Μίλησε σύντομα και ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για τις επιπτώσεις της νομοθεσίας που συζητείτε σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χορήγηση ασύλου στην Ευρώπη. Όπως και η Μελίτα, θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ στις επιπτώσεις. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι δημοσιογράφοι. Όποιο και να είναι το θέμα, ή θέματα που αφορούν ε, ε, πολύπλοκη διαδικασία από τις Βρυκλές ή κάλυψη θεμάτων διαφθοράς ή οτιδήποτε. Όλα αυτά τα θέματα είναι τα θέματα για τα οποία μου θέτουν ερωτήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσφύγων και Εξοριστέντων. Και οποιοδήποτε θέμα, η κανόνα, η νέα νομοθεσία εμφανίζεται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο θα επηρεαστεί από αυτά τα οποία γίνονται και ποιε θα είναι οι επιπτώσει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για του δημοσιογράφου. Κάθε φορά που οι, αυτοί που λαμβάνουν τι αποφάσει. συζητούν και εκπονούν νέα νομοθεσία, όλοι οι πολίτες περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών των νέων αποφάσεων στις ζωές τους. οτιδήποτε θέμα και αναφορά η νομοθεσία, τεχνολογία, τις μεταφορές, αλλά βέβαια είναι πιο σημαντικά τα πράγματα όταν έχουμε να κάνουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα ευάλωτων ατόμων που ήρθαν εδώ για να ζητήσουν την προστασία που χρειάζεται. Όπως αναφέρθηκε Φερρυπίν, ήδη θέσπισαν οι νομοθέτες ως γενικό κανόνα ότι η πρώτη χώρα στην οποία γίνεται ε, υποβάλλεται η αίτηση ασύλου θα εξετάσει την όλη διαδικασία για να τη Τι ε, γίνεται όταν αποτυγχάνει αυτή η χώρα, ποιε είναι οι επιπτώσεις στη ζωή των ατόμων. Ίσως ε, δεν αναφέρουμε μόνο στη θεωρία, στην νομοθεσία, αλλά στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα πρέπει να έχουμε κάνει τώρα. Όλες οι χώρες μέλη επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητούν το τι γίνεται με αυτούς που επιβίωσαν μετά από βασανιστήρια. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, να, του, ε, να αρχίσει η διαδικασία χορήγησης ασύλου μετά από μία πρώτη ε, ακρόση πρέπει να έχουμε ώστε ε, να τους χορηγήσουμε την δέουσα προστασία. Είναι θέμα σημαντικό που έχει επιπτώσεις. Και εάν οι νομοθέτες συμφωνήσουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων να χορηγήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στα, άτομα που, στα άτομα που ζητούν άσυλο, ώστε να μην ε, βλάψουν την ε, νοητική τους και την σωματική τους ισορροπία και ασφάλεια. Σήμερα θα πούν το απόγευμα οι ευρωβουλευτές ότι υπάρχουν κάποια συνδικές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία αυτών των ατόμων και ένα από τα αιτήματα είναι να μπορέσουν για τον κάθε ετούντα άσυλο να εξεταστούν τη θεωρία ποιες είναι ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να ισχύσουν βάσει των προβλημάτων του καθενός. Αυτή είναι η θεωρία. αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις συνθήκες κράτησης πολλές φορές όλων αυτών των ε, ε τούντων ε, άσυλο και δεν θα πρέπει κάθε φορά να επεβαίνουν ε, τα ε, δικαστήρια για να δουν αν οι συνθήκες ε, κράτησης είναι σωστές και η ερμηνεία που δίδεται από τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι πάρα πολύ ευρεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέει η οδηγία ότι ο ετών άσυλο μπορεί να κρατηθεί για να επαληθευτούν τα στοιχεία ταυτότητάς του ή να διερευνηθούν. Σωστά φαίνεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να κρατούν τον οποιοδήποτε μπαίνει εδώ χωρίς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ταυτότητα ή χωρίς ε, διαβατήριο. Όσοι έχουν προσχωρήσει στην ε, σχετική σύμβαση λέει ότι κάθε πρόσφυγας ε, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προστατεία ακόμη αν δεν έχει μαζί του τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Για ποιο λόγο. Διότι ίσως δεν είναι, πάντα ασφαλή συνθήκε υπό τι οποίε μπορεί να ζητήσει κάποιος ε, μελλοντικός πρόσφυγας ε, ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορεί να εκδιωχθεί από την χώρα του και ε, δεν μπορεί ούτε αυτό στα μέλη της οικογένειάς του να τύχουν προστασία αν ζητήσουν ταξιδιωτικά ε, και πολλές φορές η κατάσταση επιδεινώνεται τόσο πολύ γρήγορα και είναι τόσο επικίνδυνη ώστε δεν μπορεί κανείς να περάσει από τα επίσημα, ε, τις επίσημους ε, διάβλους για να βγει από τη χώρα του. Η Σύρια αυτή τη στιγμή, Φερρυπίν. Τώρα, εάν εφαρμόζοντας αυτήν την οδηγία κάποια κράτη-μέλη αρχίζουν ε, συστηματικά να κρατούν τους ετούντες άσυλο, εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να πούμε, ακούστε, αυτή δεν ήταν η πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν συμφώνησαν για το θέμα αυτό. Είπαν ότι θα πρέπει αυτό να εφαρμόζεται σε έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά ίσως ε, έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να βλέπουμε να κρατούνται υπό κάποιες συνθήκες οι μετανάστες που νομίζουν, τέτοιους μετανάστες ότι πιστεύουμε ότι έτσι είναι η συνήθιση πρακτική. Και βεβαίω φαίνεται και κάποιο μακρινή όλη αυτή η νομοθεσία των Βρυξελών, αλλά έχει επιπτώσει. Τώρα, έτσι όπω έχουν τα πράγματα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ακόμη και τα συνόδευτα παιδιά μπορούν να, ε, σε έκτακτε συνθήκε να ε, κρατηθούν. Τώρα, όσον αφορά την ε, κράτηση των ανήλικων παιδιών, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρόσεξαν πάρα πολύ οι νομοθέτες. Μίλησα με την Άγγελα την Ριφρέα που μένει στη, Μάλπα, στη Μάλτα. Μίλησε αγγλικά και θα σας πω τι ακριβώς μου είπε για αυτά τα θέματα. Λέγομαι Μερών. Έφυγα από την Ερυθρέα για να ζω χωρίς φόβο. Ήλπιζα ότι θα με καλοδεχθεί η Ευρώπη. Πίστευα ότι θα έχω την δυνατότητα που δεν είχα στο παρελθόν να κάνω κάτι στη ζωή μου. Αλλά όταν έφτασα στη Μάλτα, χωρίς κανένα λόγο, με ε, φυλάκισαν οι αρχές Ήμουνα με 19 άλλα άτομα στο ίδιο κελί και μπορούσα κάθε μέρα μόνο να υποφεληθώ από περίπατο και ήλιο μία ώρα. Μπορείτε να πείτε, δείτε πώς ε, αλλάζουν ε, οι άνθρωποι καθημερινά. Κάποιοι όμως δεν αντέχουν. Πρέπει να βγουν έξω ό,τι και να γίνει. Κάποιοι προσπάθησαν ακόμη και να απαγχωνιστούν. Κάποιοι άλλοι έπαθαν... Ε, είχαν ψυχικά προβλήματα και χρειάστηκε να πάνε σε ψυχιατρίο. Είναι ανυπόφορο να μένει κανείς ποτέ τέτοιες συνθήκες χωρίς να ξέρετε ακριβώς. Για να μπορέσω να υπομείνω αυτήν την κατάσταση, κάθε μέρα διάβαζα τη βίβλο. Μετά από 8 μήνες έτυχα προστασίας. Είμαι ελεύθερη και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά ξέρετε, πριν να φυλακιστώ, είχα σχέδια είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, είχα πράγματα να κάνω, ήθελα να βρω μια δουλειά και να ζήσω τη ζωή μου, να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Και θα ήταν πολύ πιο εύκολο το πράγμα αν δεν είχα φυλακιστεί, αν δεν είχα κρατηθεί. Η κράτηση ήτανε, δεν ήταν απαραίτητη. Τώρα θα αρχίσω να ζω σαν πρόσφυγας. Αλλά 8 μήνες που πολέμησα για την ελευθερία μου με άλλαξε πάρα πολύ. Είμαι έξω αλλά δεν είμαι όπως στο παρελθόν. Δεν επικοινωνώ με τα άτομα όπως θα έπρεπε. Ε, αν κάνεις κάτι λανθασμένο θα σε βάλω στη φυλακή. Εγώ όμω ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπω στη φυλακή. Εκτός οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όσοι κρατώνται είναι απειλή για την ασφάλειά τους. Ακόμη και όταν την χάνεις λοιπόν προστασία είσαι διαφορετικό από του άλλου. Ε, εγώ φυλακίστηκα και φοβούμαι ότι οι άνθρωποι θα με βλέπουν σαν διαφορετικό άτομα, σαν φυλακισμένη, σαν παράνομη. Έχασα την ε, ε, εμπιστοσύνη που είχα και οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι ήρθαμε για να σώσουμε τη ζωή μας. Και μετά από μήνες, όταν σε αποφυλακίζουν και σου λένε είσαι ελεύθερη, μπορείς να μείνεις στη χώρα μου, έχεις προστασία, σου φαίνονται παράλογα όλα αυτά τα οποία υπέμεινες για το τίποτα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Θα ξεκινήσει τώρα ο γύρος των ερωτήσεων. Ποιο θα ήθελε να θέσει την πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ. Στα ελληνικά φαντάζομαι. Ε, να ξαναπώ ε, Shall I say again ε, σας πω και πάλι το όνομά μου και από πού προέρχομαι. Παρακαλώ. Ε, λοιπόν, θα μιλήσω στα ελληνικά. Ε, λέγομαι Δέλη Θανάση και εκπροσωπώ το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που είναι δημόσιο μέσο επικοινωνίας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία από το UNHCR. Ποια είναι η γνώμη της. η Ελλάδα είναι μία buffer zone τελικά. Είναι μία χώρα που έχει έναν απόλυτο μικρό αριθμό αιτήσεων, αλλά μεγάλο ως ποσοστό υπό του, επί του πληθυσμού της. Θα ήθελα επίσης να κάνω μία ερώτηση στην κυρία από το ΕΚΡΕ. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την επίσημη διακυβέρνηση της χώρας με δεδομένο το δελτίο τύπου που διαβάσαμε πρόσφατα από το, το λέω στα αγγλικά, European Grassroots Anti-Racist Movement, το οποίο κρίνει ότι ο Πρωθυπουργό κύριος Σαμαράς έχει επιδείξει δίγλωσία σχετικά με το θέμα των ναζιστών και της απαράδεκτης υποστήριξης χρυσή αυγή. Αυτό το διάβασα κατευθείαν από το ε, δελτίο τύπου που έβγαλε το ΕΓΚΑΜ που είναι όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω και τις δύο κυρίες, επαναφέροντας ένα θέμα που νομίζω ε, ότι είναι σοβαρό, τουλάχιστον ε, σε εμά στην Ελλάδα ένας αξιόλογος συνάδελφος το λέω γιατί αυτός το έφερε, ο Αποστόλης ο Φωτιάδης, σε συνεργασία με συνάδελφο από τη Βαρσοβία και το Frontex, έθεσε το θέμα του Euroshoot και του συστήματος Entry-Exit, ποια είναι η θέση της ΥΠΑ ε, της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες ε, σε αυτό το δυναμικό μέτρο, το EuroSuit. Φαντάζομαι γνωρίζετε πώς πρόκειται να υλοποιηθεί. Ε, ποια είναι η θέση, αν θα διευκολύνει ή αν θα δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στο να έχουν τη δυνατότητα πραγματικοί πρόσφυγες και άνθρωποι που χρειάζονται ανθρωπιστικό καθεστώς, αν θα έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να υποβάλουν αντίστοιχες αιτήσει στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, Η Μελίτα πρώτα. Ο αριθμός των προσφύγων και αιτήσει ασύλου. Αν τα δείτε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα δείτε ότι πάντα υπάρχουν διακοιμάσεις σε κάθε χώρα. Υπάρχουν ε, ε, χώρες που ήταν κυρίως χώρες υποδοχής, ε, που τώρα μειώσαν τα ποσοστά τους και άλλες έχουν ε, ανεβάσει τα ποσοστά τους. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά εκτεθειμένη σε μια περιοχή που έχει βιώσει αρκετές κρίσεις και έχουν φύγει πολλοί από τις χώρες αυτές. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στην Ελλάδα. Αλλά στο τέλο, όπω εξηγήθηκε και από το προηγούμενο πάνελ, η Ελλάδα δεν είναι η βασική χώρα υποδοχής ε, των ετούντων άσυλο και αν το σύστημα ε, στηθεί και λειτουργεί αποτελεσματικά, τότε λογικά η χώρα θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον αριθμό των ετούντων ασύλο που φτάνουν στη χώρα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε μόνο από πλευρά αριθμού ετούν τον άσυλο, αλλά και από πλευρά δυνατοτήτω του συστήματο ασύλου να το αντιμετωπίσει και αν βελτιωθεί, φαντάζομαι ότι θα μειωθούν και οι πιέσει προ την Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα το Eurosuit, δεν έχουμε δει και πολλά πράγματα και επομένως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πώς θα λειτουργήσει ακόμα η βασική προτεραιότητα για μας, για οποιαδήποτε έλεγχο στα σύνορα, είναι ότι ο έλεγχος στα σύνορα θα πρέπει να είναι ασφαλής, ε, είναι δικαίωμα τη κάθε χώρα βέβαια να έχει ασφαλή σύνορα, αλλά δεν θα πρέπει να σφραγίζονται, να κλείνονται. Θα πρέπει πάντα να υπάρχουν διαδικασίε που θα επιτρέπουν στους ανθρώπου που αναζητούν προστασία να κάνουν αίτηση, να εξετάζεται και να καθορίζεται αν αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται γέννη προστασία και τότε θα πρέπει να γίνονται δεκτοί και στη χώρα, αλλά να ξεκινά και η διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορούμε ήδη από τα σύνορα να γνωρίζουμε ε, ε, διότι, τι γίνεται, διότι είναι πολύ δύσκολο αφενός να είναι ασφαλή τα σύνορα και να ξέρουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τη χώρα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αρνηθούμε προστασία στους ανθρώπους που χρειάζονται προστασία. Θα σχολιάσουμε όταν θα έχουμε δει περισσότερα για τη λειτουργία του συστήματος. Ευχαριστώ. Η Άννα. Απλώς να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες αιτήσει αίτησης ασύλου στην Ελλάδα ήμουν πρόσφατα και είδα ότι στους δρόμους κυκλοφορούν Αφγανοί, Πακιστανοί, Σομαλοί. Δεν υπάρχουν όμως στατιστικές, αλλά είναι πρόσφυγες. Από τη στιγμή που θέλουν να αποφύγουν κάτι το πολύ μεγάλο, κάτι πιο μεγάλο κακό που μπορεί να συμβεί στη χώρα τους και φεύγουν, θεωρούμε ότι είναι πρόσφυγες. Και όταν κάποιος πολλές φορές προσπαθήσουν να ζητήσουν άσυλο, βλέπουμε ότι δεν ε, καταλήγουν. Και λένε, ακόμη και αν ζητήσουμε χαρτιά, τι θα κερδίσουμε. Τίποτε δεν ε, κερδίζουν αυτοί που τα έχουν και χάνουν την πίστη τους. Αν λοιπόν ε, κάποιος χάσει την πίστη του γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα, είναι άσχημα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά άτομα που υπάρχουν εκεί που χρειάζονται προστασία και το σύστημα δεν είναι ε, σε θέση να τους εντοπίσει, να τους ταυτοποιήσει και να τους προστατεύσει. Βεβαίως, είναι πολύπλοκη κατάσταση. Πολλά πράγματα συνέβησαν συγχρόνως. Έχουμε μαζικές ε, εισρωές τέτοιου είδους ατόμων για χρόνια και εξαιτία της ε, ε, γεωγραφικής θέσης, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη πολιτική. Ίσως και σήμερα υπάρχουν πολλά προβλήματα με πολλά άτομα και όλοι όταν αρχίζουν τα προβλήματα αρχίζει να δείχνει το λάθος στον άλλο. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για την πολιτική για το τι είπε ο Α ή Β πολιτικός. Αλλά βλέπουμε στην Ελλάδα ότι πολλά άτομα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν τους άλλους. Και είναι κρίμα, θα ήταν κρίμα η, η εικόνα της χώρας να αμαυρώνεται από την Χρυσή Αυγή και αυτούς που κάνουν πράγματα αρνητικά, ενώ υπάρχουν πολλοί που κάνουν τόσα θετικά και βοηθούν τόσο πολύ. Και θα πρέπει να σκεφτούμε του πάντε. και να μην είμαστε πολύ απεσιόδοξοι. Για το σου εγώ δεν είμαι ειδική για το φάκελο αυτό, αλλά όπω είπε η Μελίτα, οι συνοριακοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται με εξισορροπημένο τρόπο. Βεβαίω θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν οι χώρε ποιον θέλουν ναι ή όχι, αλλά αυτό δεν είναι σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται ενάντια στα θεμελιώδη δικαιώματα του οποιοδήποτε ή του κάθε ε, ετούντα άσυλο. Βεβαίως, εάν υπάρχουν εξωτερικά ε, σύνορα και συμβαίνουν πράγματα εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντό των εσωτερικών σύνορων, είμαστε κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνοι. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Με ακούτε? YouTube Samanda. Αυστρικά μέσα ενημέρωσης. Είπατε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ε, ε, διαφορές όσον αφορά τα ποσοστά χωρίς προσφύγων στην Ευρώπη. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γενικά ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε τέτοιες μεγάλες διαφορές. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι νέες οδηγίες θα βελτιώσουν την ε, κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να ευρεθεί η χρυσή τομή. Η επόμενη ερώτηση αφορά το Eurodac. Και στις δύο μιλήτριες. Κατά την άποψή σας, Ποιο είναι το πιο προβληματικό θέμα για την πρακτική εφαρμογή του Eurodac. Βλέπουμε διαφορές σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είπα προηγουμένως. Το να έχουμε κανόνες και τις οδηγίες. Είχαμε και στο παρελθόν οδηγίες. Δεν αρχίζουμε με το κοινό σύστημα χορηγής ασύλου εκ του μηδενός το να ε, έχουμε στη θεωρία του κανόνε και να του εφαρμόσουμε στην πράξη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση. Η Άννα επίση είπε ότι μπορείτε να έχετε ένα σύνολο κανόνων, αλλά το θέμα είναι πώ θα ερμηνευτούν. Η ερμηνεία των κανόνων είναι σημαντικό θέμα. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία συζητώνται σε αυτό το τομέα και σε θέματα εσωτερικής νομοθεσίας και η στάση όλων των πολιτών προς τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν Πακιστανούς, ε, Αφγανούς που ζητούν ε, άσυλο και όπως λένε κάποιοι είναι λαχείο η προστασία τη χώρα. Και τώρα είμαστε σε αυτή την κρίσιμη φάση. Έχουμε επί χάρτου τη θεωρία, αλλά θα πρέπει και τους κανόνες, αλλά θα πρέπει να τους θέσουμε σε εφαρμογή και να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το Eurodac. Ναι, το Eurodac. Αυτό το οποίο μας απασχολεί με το Eurodac είναι το εξής. Ε, ασκήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις ώστε να μπορέσουν να είναι στη διάθεση των διοκτικών αρχών τα στοιχεία του Eurodac. Είμαστε αντίθετοι, χάσαμε τη μάχη όμως. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συνθήκε προστασίας και ασφαλείας. Τι κάνει ένας αστυνομικός ο οποίος ερευνά μία περίσταση όταν ε, έχει τα δεδομένα μπροστά του για ε, κάποιον ερευνά όλα αυτά τα, τα στοιχεία και να μοιραστεί τις πληροφορίες με την χώρα καταγωγής είναι προνόμιο των αστυνομικών και εθνικών διοκτικών αρχών. Αλλά για τους πρόσφυγες δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους συνεργασία με την χώρα καταγωγής διότι τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο το άτομο που ζητά ασύλο, αλλά και όλο το οικογενειακό του περιβάλλον. Και βλέπουμε εδώ διαφορές. Έχουν υπάρξει σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι συνθήκες ε, προστασίας και ασφαλεία και οι δικλείδε σχετικές, αλλά σε άλλες περιπτώσεις όχι. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να είναι στη διάθεση των υπεύθυνων αρχών για την χορήγηση του ασύλου και όχι για όλες τις διοκτικές αρχές και τις αρχές επιβολής νόμου. Αλλά τη χάσαμε αυτή τη μάχη και προσπαθούμε λοιπόν αυτές τις συνθήκες προστασίας και ασφαλείας να είναι οι καλύτερες δυνατές ώστε να αποτρέπεται η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής εις βάρος των ατόμων που είναι πρόσφυγες ζητούν άσυλο. Για το Eurodac συμφωνώ απόλυτα. Το γεγονό ότι θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τους αιτήντες άσυλο ορισμένες φορές να φτάσουν τα στοιχεία τους στη χώρα καταγωγή του. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να ανησυχούν ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να φτάσουν στη χώρα τους, μπορεί να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που φοβούνται θα προσπαθήσουν να αποφύγουν το σύστημα και να προσπαθήσουν να το παρακάμψουν. Ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο στη θεωρία θα έπρεπε να διευκολύνει την προστασία τους μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα και αυτό φυσικά είναι κίνδυνος και να μην ξεχνούμε και το θέμα του στίγματος, ε, γιατί εξετάζουμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Ευρω... Τα στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών ε, δεν εξετάζουν ε, στοιχεία σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας. Γιατί λοιπόν οι αιτούντες ίσολων να ε, τους αντιμετωπίζουμε ως εγκληματίες. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που μας ανησυχούν. Όσον αφορά τώρα το Δουβλίνο και το Eurodac μαζί. Στο Δουβλίνο υπάρχει μία σειρά από κριτήρια ιεραρχημένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι κατά πόσον κάποιος διαθέτει οικογένεια στις χώρες αυτές και μας υπενθύμησαν ότι αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά με αρκετούς εταίρους σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουμε πώς ε, λειτουργεί αυτό στην πράξη. Ο γενικός κανένας στην πράξη είναι ότι η πρώτη χώρα ε, εισόδου είναι αυτός, ε, αυτή η οποία ισχύει, διότι ε, μέσω του γύροντα υπάρχει ένα hit και βρίσκουμε σε ποια χώρα πήγες και ε, δεν κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να εντοπίσουν τα μέλη της οικογένειας κάποιου. Ωραία. Φτάνουμε προς το τέλος. Ξαφνικά βλέπω ότι έχουμε ε, σωρία ερωτήσεων. Τρεις ε, ενετόπισα που θέλουν να θέσουν ερώτηση. Θα σταματήσουμε μετά από αυτούς τους τρεις και θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε σύντομοι στο προκείμενο και σας παρακαλώ να απαντήσετε και σύντομα ο κύριος εκεί στο βάθος καταρχάς. Ευχαριστώ. Τζουζέπε Ντιμίκο από την Κατσέτα Τελμετζορτζόρνο θα ήθελα να ρωτήσω στην κυρία Λόπες Φοντάνα εάν η επιστολή που μας διαβάσατε ε, έχει επαληθευτεί και αν έχει διαβιβαστεί στους αρμοδίους για να δούμε ε, να δουν μάλλον οι αρχές αν ε, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο και αν υπάρχει αντίστοιχη ε, περίπτωση και σε άλλες χώρες. Η συγκεκριμένη επιστολή είναι συνέχεια μιας ιδιωτικής συζήτησης που είχα εγώ με τη συγκεκριμένη κοπέλα ε, εγώ τη το ζήτησα να το γράψει γιατί ήξερα ότι θα μεταδοθεί ζωντανή, αλλά αυτό το, το θέμα δεν είναι καινούριο. Γνωρίζουμε τις συνθήκες κράτησης ε, των προσφύγων. Στη Μάλτα είναι ε, ακόμα πιο επωνίδεστες οι συνθήκες, διότι είναι πολύ μακρά η διαδικασία. Όποιος φτάνει κρατείται, μόνο ανήλικοι και τα άτομα απελευθερώνονται. Υπάρχει λοιπόν η επιστολή, μπορείτε να τη διαβιβάσετε σε όλο τον κόσμο, αλλά οι συνθήκες κράτησης είναι γνωστές στη σπάση νομίζω και το ξέρουν όλοι ότι αυτό συμβαίνει. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και η πατιαρμοστία για του πρόσφυγε προσπαθούν να αλλάξουν το θέμα των συνθήκων κράτηση, γιατί γνωρίζουμε ότι οι αρχέ πρέπει να ελέγχουν ε, ποιο βρίσκεται στη χώρα και ποιοι είναι οι αιτούντε άσυλο, αλλά υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Και πάντα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία των ανθρώπων, ε, τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο ελπίζουμε ότι θα πείσει κάποιες κυβερνήσεις. Οι συνθήκες, ε, οι εναλλακτικές λύσεις κράτησης είναι φθηνότερες από την κράτηση. Ο κύριος Στοβάθος, Ευχαριστώ. Αμέτ Τζεμάη, δημοσιογράφος από τη Media Press ε, στη Γαλλία. Θα ήθελα να σας θέσω τρεις ερωτήσεις υπό την έννοια παρατήρησης. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους ετούντες άσυλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ αυτού που θα μπορούσε να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή τι ψηφίζουν οι ευρωβουλευτέ και ε, την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου στις χώρες. Για να γνωρίζετε λίγο τι συμβαίνει στη Γαλλία, γνωρίζω ότι συχνά οι δύο αστυνομικέ αρχές δεν σέβονται την νομοθεσία και όταν μιλάτε για την κράτηση νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περίπτωση. Η ερώτησή μου είναι η εξής οι οργανώσεις που εκπροσωπείτε εσεί. Και δεδομένου του σημασία στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσαμε να έχουμε ίσω και κάποιε εκστρατείε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε τρει βασικέ ε, συνιστώσει. Οι ευρωβουλευτέ, ε, διότι μπορεί να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτέ ένα νόμο εδώ, αλλά όταν βρίσκονται στην περιφέρειά του ε, επηρεάζονται λίγο από την κοινή γνώμη και μπορεί να αλλάξουν πρακτική. Δεύτερη συνιστόσα, ε, κατευθυνόμενη προς την κοινό γνώμη. Ε, η συνάδελφος από την Ελλάδα το ανέφερε προηγουμένως. Γνωρίζουμε ότι η επικυρότητα, ε, ιδίω όσον αφορά τους ετούντες άσυλο στην Ελλάδα, στη Μάλτα και αλλού, ε, είναι πολύ δραματική, διότι έχουμε υπάρξει μάρτυρες ε, βιαιοτήτων ε, εκ μέρους συγκεκριμένων πολιτών κατά ετούντων άσυλο. Και μια τρίτη δράση να απευθυνθούμε κυρίως ε, στις αστυνομικές διευθύνσεις που είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και αν δεν κάνω λάθος η νομοθεσία που ψηφίζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερτερεί της εθνικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα αγγλικά. αναφέρεστε σε αυτό το οποίο είπε και η Άννα και εγώ. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι η θεωρία και διαφορετική η πρακτική. Προσπαθούμε λοιπόν σήμερα να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική κουλτούρα. Και όλα αυτά, στις, στοχευμένες ομάδες για τις οποίες μιλήσατε προσπαθούμε μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, είπα της αρμοστίας, ε, δικηγόρων και άλλων φορέων να δούμε πώς θα, συζητώντας το όλο θέμα, θα συντονιστούμε. Όσον αφορά τις ε, εκστρατείες ε, για να μπορέσει να αφυπνιστεί η, δι... Ε, η κοινή γνώμη. Πολλά γίνονται. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα γίνονται τέτοιου είδους εκστρατείες που υποστηρίζουν πολλοί φορείς. Διανούμενοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες. Και δεν είναι κάτι το οποίο κατευθύνεται από τα Ηνωμένα Έθνη, γίνεται και από τους, ε, το γκλήρο μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα κτλ. Τώρα, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης ακόμη και των αστυνομικών. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, υπάρχει ως πρόγραμμα, αλλά σωστά δεν είναι επαρκή όλα αυτά. Πρέπει να ενεργήσουμε περισσότερο, γιατί όσο περισσότερο απομακρύνεται κανείς από τα θεσμικά όργανα και τις Βρυξέλλες, όλο περισσότερο οι πάντες επηρεάζονται από το τι πιστεύει η κοινή γνώμη για τα θέματα της προστασίας των προσφύγων που πρέπει να εξασφαλίσουμε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, η αρμοστία, οι διανοούμενοι, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να μπορέσουν να αφυπνήσουν την κοινή γνώμη για τα θέματα καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κάτι που γνωρίζει η Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες συμβαίνουν κάποια πράγματα. Γιατί, Γιατί πολλές φορές ε, οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που θέτουν τον... Ε, που κάνουν την προειδοποίηση για να αφυπνίσει και το κάτι δεν πάει καλά. Ευχαριστώ. Θέλει Κάποια άλλη συμμετέχουσα να κάνει μια ερώτηση. Καμαρέρα. Από την Βαρκελόνη. Τι συμβαίνει με αυτούς οι οποίοι έρχονται από την περιοχή του Καυκάσου και τη Ρωσία και ζητούν άσυλο. Πρόκειται για πολλά άτομα που έχουν ειδικά προβλήματα πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την όλη πολιτική. Δεν θα πρέπει το άσυλο να το συγχαίουμε με την ε, πολιτική χρειά του όλου προβλήματος και με τις σχέσεις μεταξύ ε, κρατών, χώρα καταγωγής, χώρα υποδοχής. Στη θεωρία. Αυτή είναι η θεωρία. Τώρα στην πράξη. έχουμε δει να υπάρχουν προβλήματα και πολλές φορές την όλη ζήτηση την επηρεάζουν και διάφορες ε, οικονομικές, ε, οικονομικού τύπου προσεγγίσεις και απόψεις. Τώρα, εγώ δεν έχω στατιστικές τώρα, αλλά πόσον ξέρω, η δυνατότητα που έχει ένας Ρώσος, ένας Τσετσένος από τον Κάφκασο, τέλος πάντων, να τύχει προστασίας, είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με τη χώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά για την Πολωνία, πολύ υψηλά για την Αυστρία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Που και πάλι, τι καταδεικνύουν. Ότι επί χάρτου η εναρμόνιση δεν επαρκεί. Το επόμενο βήμα θα είναι στο επίπεδο εφαρμογής να έχουμε εναρμονισμένο τρόπο ε, πρακτικής ε, της χορήγησης αυτού του λαχείου που λέγεται άσυλο. Ε, εμείς έχουμε μία ομάδα που είναι η εξειδικευμένη για τα άτομα που ε, πρόχνονται από την ε, ε, Ρωσία. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε αργότερα αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας, κυρίως τα μέλη του πάνελ. Όπως ξέρετε, προβλέπετε στον πέμπτο όροφο μία εκδήλωση για σας έναν όροφο επάνω. Είμαστε στον τέταρτο, δηλαδή να πάμε στον πέμπτο όροφο. Θα έρθετε κι εσείς παρακαλώ. Μπορώ. Και μην ξεχνάτε ότι ξαναρχίζουμε στις δύο ακριβώς με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Άννα θέλει να πει κάτι σύντομα. Όσοι μένουν έως αύριο, είδα ότι πολλοί ενδιαφέρονται για τον κανονισμό του Δουβλίνου και πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Εδώ στο Κοινοβούλιο, σήμερα το πρωί, έχουμε μία εκδήλωση για το Dublin, δηλαδή κάναμε μία μελέτη για να δούμε πώς λειτουργεί ο κανονισμός στις διάφορες χώρες. Δηλαδή, από τη θεωρία στην πράξη. Τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και θα έρθουν πολλά άτομα, ειδικά που θα μας μιλήσουν για αυτό το θέμα και οι συγκητέ που, ε, που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις θα συζητήσουν το όλο θέμα αύριο. Αν θέλετε και είστε εδώ μπορείτε να συμμετάσχετε. Λεπτομέρειες πώς μπορούμε να πάμε, πού θα γίνει η συνάντηση αυτή. Ναι, ναι. Όταν έχω τα στοιχεία θα σας τα δώσουμε. Λοιπόν, στον πέμπτο όροφο. Αμέσως για τη ρεσεψιόν. Thank you.